bonjour à tous. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε Άρχεται η συνεδρίαση. Θα κάνω πρώτα μια ανακοίνωση. Έλαβα από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αιτήσεις διορισμού στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Ο κατάλογος αυτών των διορισμών θα περιληφθεί στα πρακτικά αυτή τη συνεδρίασης και αν δεν έχουν υποβληθεί παρατηρήσεις μέχρι την έγκριση των πρακτικών, αυτοί οι διορισμοί θα θεωρηθούν ως εγκριθέντες. Τώρα έχουμε την... Τα του Δικού Συμβουλίου Εκοφήν τη 7η Σεπτεμβρίου και τη Δηλώσει Συμβουλίου και τη Επιτροπή. Εξ ονόματο του Συμβουλίου θα δώσω πρώτα το λόγο στον Υπουργό Οικονομικών του Βελγίου, τον κύριο Ρέντερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ απλά θα ήθελα να σας πω τη συνεδρίαση του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες μας επέτρεψε να σημειώσουμε πρόοδο σε δύο φακέλους εγκρίνοντας το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο στα πλαίσια τη ε, δημοσιονομική εξυγίανση και την άλλη διαδικασία παρακολούθηση του προπολογισμού, επιβεβαιώνοντα επίση την συμφωνία η οποία είχε γίνει στην τριμερή συνάντηση μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπή για το σύνολο των κειμένων που αφορούν την χρηματοπιστωτική εποπτεία. Είχαμε δύο συζητήσει επίση που θα συνεχιστούν στη διάρκεια αυτού του μήνα στο ε, άτυπο ΕΚΟΦΗΝ με σκοπό να προοδεύσουμε στη διάρκεια του εξαμήνου για την ε, τραπεζική συμβολή και για την ε, πρώτον και δεύτερον την επιβολή φόρων στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Για το πρώτο εξάμεινο αυτή θα είναι ένα πρώτο στάδιο που θα μας επιτρέψει κατόπιν του χρόνου να ξεκινήσουμε την νέα δημοσιονομική διαδικασία με την Επιτροπή ζητώντα από την άνοιξη στις χώρες να μας υποβάλουν δημοσιονομικά στοιχεία τις μεγάλες κατευθύνσεις του προϋπολογισμού τους χωρίς βεβαίως λεπτομέρειες για κάθε κονδύλι προτού συνεχιστεί αυτή η διαδικασία με την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να προσθέσουμε νέες διατάξεις κυρίως που θα αφορούν κυρώσεις. Η Προεδρία θα προσπαθήσει ε, να, εφαρμόσει αυτές τις κυρώσεις με, σε συνεργασία με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπό την ε, εποπτεία του αρμόδιου επιτρόπου. Θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές και όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έλαβαν μέρος σε αυτή τη αναζήτηση συνένεσης για τα διάφορα κείμενα και τον Επίτροπο Μπερνιέ και τους συνεργάτες του και την Ισπανική και τη Σουηδική Προεδρία που προηγήθηκαν ήταν ώστε πλέον σήμερα να έχουμε ένα κείμενο και κείμενα μάλλον που από την 1η Ιανουαρίου θα μας επιτρέψουν να εφαρμόσουμε τα νέες διαδικασίες εποπτείες, παρακολούθησης και την Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου ώστε να δημιουργήσουμε μια νέα αρχιτεκτονική για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την εποπτεία του. Αυτό δεν είναι το τελικό στάδιο, αλλά η έναρξη, η έναρξη μια, ενός νέου, ε, μιας νέας ευρωπαϊκής οργάνωσης και θα ακολουθήσουν πάρα πολλές συζητήσεις που θα μας επιτρέψουν να εγκρίνουμε διάφορα κείμενα τα οποία θα έχει την ευκαιρία με την πάρα των εβδομάδων να σας παρουσιάζει ο Μισελ Μπερνιέ. Θα τηρήσουμε ένα πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα για το θέμα αυτό. Αυτά για τα δύο σημεία που αποτέλεσαν αντικείμενο επίσημων αποφάσεων του ΕΚΟΦΗΝ. Είχαμε, όπως σας είπα, και συζητήσεις για δύο άλλα θέματα. Τραπεζική συμβολή και η επιβολή ε, φόρων στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Σε ό,τι αφορά την τραπεζική εισφορά, η συζήτηση στο ΕΚΟΦΗΝ μας επέτρεψε να ε, προσδιορίσουμε ορισμένες κατευθύνσεις και ε, οπότε θα μπορέσει να μας υποβάλει πιο συγκεκριμένες προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει, όπω κάναμε για την ε, εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματο, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση του επόμενου μήνε, καταλήγοντα σε μηχανισμού που θα επιτρέψουν ουσιαστικό συντονισμό στην Ευρώπη. Ορισμένε χώρε ήδη ε, ε κάνουν ορισμένε παρακρατήσει σε, σε ό,τι αφορά το, το τραπεζικό τομέα, αλλά όλα αυτά θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξανασυζητούσαμε στη διάρκεια του άτυπου συμβουλίου αυτού του μήνα. Τώρα, για την επιβολή φόρων στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Η συζήτηση ήταν πολύ πιο ζωηρή. Δεν έχουμε ακόμα καταλήξει σε συνένεση, κάτι που είναι φυσικό. Ήταν μια πρώτη ουσιαστική συζήτηση είχαμε τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε τα θέματα που πρέπει να ε, ληφθούν υπόψη για την επιβολή ε, μιας τέτοιας φορολογίας και κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να υπάρξουν και συζητήσεις με άλλους εταίρους στο G20 θα έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε με τους εταίρους των αναδιωμένων χωρών και ε, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού θα γίνουν πολλές προσπάθειες για να πιστούν όλοι και μετά θα χρειαστεί να γίνουν επιλογές κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί και αν, με τέτοια φορολογία και πού θα πηγαίνουν και ποιος, πού θα διοχετεύονται τα έσοδα, αυτά τα φορολογικά έσοδα. Ορισμένοι ε, επιμένουν ότι αυτό πρέπει να ε, γίνει για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και για την καταπολέμηση της ε, κλιματικής αλλαγής. Αυτά είχα να σας πω, κυρία Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο Μπαρνιέ για την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές και εγώ θα ήθελα με τη σειρά μου να σας πω λίγα λόγια ως προς την προσέγγιση μας ε, για το ΕΚΟΦΗΝ, εξ ονόματος του Όλη Ρεν και του Επιτρόπου Σεμέτα. Υπάρχουν τέσσερα σημεία που, όπως είπε και ο Βέλγος Υπουργός, ε, διέκριναν αυτό το Συμβούλιο. Επειδή το Κοινοβούλιο συμμετείχε σε αυτές τις διαδικασίες και έθεσε ένα μείζον ζήτημα δομικού χαρακτήρα που με απασχόλησε επί μακρόν, από τότε που μας αναθέσατε αυτό το έργο το Φεβρουάριο είναι το θέμα της εποπτείας, διότι η εποπτεία είναι ύψης της σημασίας και πλαισιώνει το ολοοικοδόμημα έτσι ώστε να μπορέσουμε κομμάτι-κομμάτι να εφαρμόσουμε αυτά τα ε, δεδομένα της ε, κρίσης, δηλαδή να έχουμε μια ευφυή ε, εποπτεία και ρύθμιση και να μας ανοίξει το δρόμο έτσι ώστε κανένα προϊόν, καμία ε, αγορά και καμία χρηματοπιστωτική, κανένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα να μην ξεφύγει από αυτή τη ρύθμιση. Πιστεύω ότι σε μερικές εβδομάδες και το Κοινοβούλιο ε, θα ε, Εγκρίνω αυτό το πλαίσιο οι ε, κύριοι Σκίνερ, Σάντσες ε, και πολλοί άλλοι, μεταξύ των οποίων και η Σάρον Μπόουλς, ε, εμψύχωσαν αυτόν τον τριμερή διάλογο στα πλαίσια της ε, Βελγικής Προεδρίας, μέσα στα πλαίσια μιας εκούσιας συμφωνίας, διαδικασία που άρχισε υπό την Σουηδική και Ισπανική Προεδρία. Ο βασικός λόγος της πρότασης της Επιτροπής για την εποπτεία είναι η πολύ σημαντική εργασία του Ζακ Ντελαροζιέρ για να φτάσουμε στα πρώτα δεδομένα απότοκα της κρίσης. Από τον Ιανουάριο η Κομισιόν θα, θα ε, εποπτεύσει αυτές τις τρεις αρχές, καταρχήν το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου και θα προβάλλει όλους τους ε, ελέγχους που επιβάλλονται, διότι στο ίμιση των χωρών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ίμιση των τραπεζών, ανήκουν σε άλλες χώρες. Πρόκειται για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν διεθνικό χαρακτήρα. Άρα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους ε, συστημικούς κινδύνους που απορρέουν από αυτή την κατάσταση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Προεδρία και τους δικούς σας εισηγητές για τη σημαντική αυτή εργασία, για την επιτυχία των, ε, του πρώτου αυτού, αυτού βήματος, όπως είπε και ο κύριος Ρέιντερς. Και ήδη την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσω για τη ρύθμιση των παραγόγων, τις ανοιχτές πωλήσει και τα ιδρύματα επιστοληπτικής ικανότητας, στους οργανισμούς επιστοληπτικής ικανότητας έτσι ώστε θα δούμε πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε για μια ε, φορολόγηση. Η Βελγική Προεδρία είπε ότι δεν πρέπει να συγχαίουμε τα δύο ζητήματα τα οποία είναι διαφορετικά. Ως προς τη χρηματοδότηση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ως προς αυτό το Ταμείο Εξυγίανσης. Είναι μια ε, διαδικασία που άρχισε στο Συμβούλιο. Η συζήτηση είναι πολύ χρήσιμη διότι από αυτό το γύρο του τραπεζιού βλέπουμε λίγο σαφέστερα την κατάσταση. Στη Μαδρίτη, στο άτυπο συμβούλιο, μίλησα για μια ε, εργαλειοθήκη έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την ε, κρίση γιατί η πρόληψη στοιχίζει πολύ λιγότερο από τη θεραπεία. Αυτό αφορά για όλους ε, τους τομείς, μεταξύ των οποίων και την χρηματοπιστωτική κρίση. Ο φορολογούμενος δεν πρέπει να βρίσκεται στην εμπροστοφυλακή. Θα πρέπει οι τράπεζες να καταβάλουν το αντίτιμο. Μιλήσαμε λοιπόν για μια εργαλειοθήκη μεταξύ αυτών των, των, στοιχείων μάλλον που την απαρτίζουν είναι και το Ταμείο Εξυγίανσης. Η κυρία Φερέιρα ε, επιτέλεσε αυτό το έργο εξ ονόματός σας και τον Οκτώβριο θα προβώ σε μία ανακοίνωση με βάση τα δεδομένα της κυρίας Φερέιρα στο Συμβούλιο Υπουργών, διότι τον Οκτώβριο θα έχουμε προχωρήσει σε μια σημαντική διαδικασία, τη διαδικασία της Βασιλείας, ως προς την κεφαλαιοποίηση ιδίων πόρων. Και όταν μιλάμε για συνεισφορά, η εισφορά των τραπεζών θα πρέπει να ε, στοιχειοθετήσουμε όλα τα δεδομένα, να έχουμε δηλαδή μία οριοθέτηση έτσι ώστε να μην ξεφύγει κανένας, να μην, έχουμε, ε, να μην ισχύει το ρητό business as usual να δούμε πώς λειτουργεί η οικονομία σορευτικά και πώς λειτουργούν σορευτικά όλα αυτά τα μέτρα. Γι' αυτό θα προβώ σε μια ανακοίνωση τον Οκτώβριο για την πρόληψη μελλοντικών κρίσεων και την ευθύνη που φέρουν οι τράπεζες, καθώς και το Ταμείο Εξυγίανσης, γιατί η Γερμανία και η Σουηδία έχουν θέσει αυτή την ιδέα επιτάπητος. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα συντονισμένο σύστημα με έναν κοινό κόρμο έτσι ώστε να μην υπάρχει κακός ε, νοούμενος συντονισμός και διπλή φορολογία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Όπως είπε ο κύριος Ράιντερς, τα δεδομένα, η φορολόγηση μάλλον των συναλλαγών, των παγκοσμίων συναλλαγών έχει αρχίσει σε επίπεδο G20. Δεν ήταν όλοι ιδιαίτερα ενθουσιώδεις Πολλοί πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές μπορούν να συνεισφέρουν στην χρηματοδότηση αυτής της μεγάλης πρόκλησης έτσι ώστε ο κόσμος να είναι πιο δίκαιος πιο και πιο σταθερός. Άρα θα πρέπει να είναι πιο δίκαιος, κάτι το οποίο δεν ισχύει σήμερα. Θα πρέπει να δούμε τις κλιματικές αλλαγές, ε, τα διατροφικά δεδομένα, την κρίση, το περιβάλλον και να αντιμετωπίσουμε τις φτωχότερες χώρες. Άρα θα πρέπει να ε, επικρατήσει η αρχή της δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει πάντα συνένεση στο Συμβούλιο Υπουργών. Ο συνάδελφος Σεμέτα υπέβαλε ε, μία πρώτη ανακοίνωση, ένα πρώτο υπόμνημα και θα ξαναδούμε την φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπως προβλέπεται τον Οκτώβριο. Δεν θα ήθελα να ε, επαναλάβω αυτά που είπε ο κύριος Ράιντερ σε σχέση με τη σταθερότητα ως προς τον τομέα της σύγκλησης. Έχει συσταθεί μια task force και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα επιτρέψει μια δημοσιονομική ανάλυση όλων των χωρών μέσα στα πλαίσια της εθνικής κυριαρχίας. Θα έχουμε όμως μια φωτογράφηση, μια ανείχνευση της ε, ευρωπαϊκής κατάστασης σε σχέση με την οικονομική της πολιτική. Το Συμβούλιο θα εργαστεί με βάση και τις εκθέσεις της Επιτροπής επί του θέματος. Κατά το γεύμα, ο Ντίντια Ράιντερς προέβαλε δύο συζητήσεις. Η μία μας αφορά. Αφορά το EASB, δηλαδή τον Διεθνή Οργανισμό Λογιστικών Προτύπων, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διάβια και ήδη είπα στην Προεδρία ότι στο άτυπο Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου θα υποβάλω μία έκθεση που αφορά και το Κοινοβούλιο σε σχέση με την διατλαντική ρύθμιση. Στις, στους G20 δεν είμαστε οι μόνοι. Δεν είμαστε μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών μόνο. Θα πρέπει να εποπτεύουμε τα παράλληλα μέτρα τα οποία εξήγηλε και ο πρόεδρος Ομπάμα στο Αμερικανικό Κογκρέσο σε σχέση με την εποπτεία και τη ρύθμιση. Άρα ε, προβαίνω σε μια συγκριτική μελέτη για το τι γίνεται στη ΣΥΠΑ αυτή τη στιγμή και τι κάνουμε εμείς στην Ευρώπη για να έχουμε μια παράλληλη πορεία και να φτάσουμε στους ίδιους στόχους με παρόμοια μέτρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε και θα δώσω τώρα το λόγο στους ομιλητές των ομάδων ξεκινώντας με την κυρία Βοντονόλ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα ήθελα να σας πω ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ για τη συμφωνία που ε, επιτευχθεί για ευρωπαϊκή εποπτεία των τραπεζών. Είναι σημαντικό ορόσημο Ορισμένα κράτη-μέλη στην αρχή εργούσαν ε, και εμπόδιζαν τις διαδικασίες, αλλά οι δικοί μας οι ε, ε, επέμεναν και με την επιμονή και τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Βελγικής Προεδρίας προχωρήσαμε. Είναι πολύ σημαντικά τα βήματα. Θα πρέπει να ενισχυθεί η οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης. Συζητήσατε στο ΕΚΟΦΗΝ και για τους διαφόρους φόρους ε, με τους οποίους θα επιβαρυνθούν οι τράπεζες, γιατί θα πρέπει και εκείνες να υπομισθούν το κόστος της κρίσης. Λέτε για το G20, αλλά η πρόοδος που έχει γίνει είναι μικρή. Γι' αυτό συμφωνεί με τα συμπεράσματα και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που λέγουν ότι αν δεν επιτύχει αυτό διεθνώς, μπορούμε εμείς στην Ευρώπη να αναλάβουμε ε, πρωτοβουλία και να δείξουμε ηγετική στάση και να εισαγάγουμε ένα είδος ε, τραπεζικού τέλους ή τραπεζικού φόρου. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει με τρόπο συντονισμένο Ορισμένα κράτη-μέλη αρχίζουν να επιβάλλουν τέτοιου φόρου, αλλά αυτό, προσοχή, είναι απειλή για την εσωτερική αγορά μας. Κύριε ε, Μπαρνιέ, παρακαλώ, ε, χρησιμοποιήστε το δικαίωμα πρωτοβουλία που έχετε για να είμαστε συντονισμένοι, στοιχημένοι και να προχωρήσουμε στην ίδια κατεύθυνση για τη φορολόγηση των τραπεζών. Και όπως και με την εποπτεία ε, θα έχετε στο πλευρό σας το κοινοβούλιο. Όταν πρόκειται τώρα για τον φόρο επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Αυτό είναι κατεξοχή κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει ακριβώς σε επίπεδο G20 και παρακαλώ πολεμήστε το, προσπαθήστε το αυτό. Θα ήθελα όμως να προειδοποιήσω και πάλι και η Ευρώπη να μην απομονωθεί, να μην προχωρεί μόνη της. θέλει να το επιβάλλει ο κύριος Σούλτ και το γνωρίζω αυτό, αλλά τα μειονεκτήματα είναι περισσότερα από τα πλεονεκτήματα, γιατί οι συναλλαγέ είναι παγκόσμια ε, οικονομική δραστηριότητα και αν το κάνει αυτό μόνη τη η Ευρώπη θα την παρακάμψουν οι ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγέ. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο κύριο Ούντο Μπούλμαν για 1,5 λεπτό. Κύριε Προεδρεύον, κύριε Επίτροπε, Συγχαρητήρια για την τραπεζική υποπτία. Το Κοινοβούλιο έκανε όλη τη δουλειά και εσείς βοηθήσατε πολύ. Γι' αυτό φτάσαμε σε ένα τόσο καλό αποτέλεσμα. Δυστυχώ όμω οφείλω να πω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε τα νέα καθήκοντα. Γιατί σε άλλα σημεία που έχουμε πολύ από μια καλή ρύθμιση. Βλέπε μάνατζερ των hedge funds, πόρο απέχει από τη λύση. Και κάνω μια έκκληση τώρα και ε, στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κινηθείτε, γιατί αν δεν κινηθείτε εσεί δεν θα υπάρξει καλή ρύθμιση. Χρειαζόμαστε ε, το ίδιο δίκαιο για όλου. Και οι μάνατζερ εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει κάποια στιγμή να υφίστανται τα ίδια και να υπόκεινται στις ίδιες ρυθμίσεις. Αλλιώς θα έχουμε μειονεκτική θέση για την Ευρώπη. Δεν θέλουμε να καταστήσουμε όμοιρο ένα ολόκληρο κλάδο της οικονομίας, αλλά να βοηθήσουμε και να ε, απομονώσουμε τα μαύρα πρόβατα. Αλλιώς δεν πρόκειται να υπάρξει καλή ρύθμιση. Και θέλω να σας προειδοποιήσω. Μην πιστεύετε σε κάποιες έτσι εύκολες νίκες επειδή θα μας διχάσετε στο κοινοβούλιο και θα περάσει το δικό σας. Όχι, όχι. γιατί ε, πιέζουν τα λόμπι και δεν θα πρέπει να γονατίσει η Ευρώπη μπροστά του. Για τι συναλλαγέ και τη φορολόγηση διαφωνώ με την κυρία Βότμαν Κόλ. Όχι, η Ευρώπη περιμένει απαντήσει. και θα πρέπει να δώσετε απαντήσει. Μην γυρίζετε πίσω από του G20 και μα πείτε άλλοι που είμαστε πάρα πολύ δεν καταφέραμε τίποτα και τώρα σταυρώνουμε τα χέρια. Όχι, θα πρέπει να δράσει η Ευρώπη, να κάνει αποφασιστικά βήματα με του Ευρωπαίου και θα το κάνουμε. Σκεφτείτε το στις διαπραγματεύσεις σας παρακαλώ στο G20. Χρειαζόμαστε απάντηση. Και αν δεν υπάρξει στο G20 ας είναι αυτή η ευρωπαϊκή. Ευχαριστώ κύριε Μπόλμαν. Η κυρία Γκούλαρ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή και την Βελγική Προεδρία που μας βοήθησαν να δημιουργήσουμε αυτό το σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο της, ε, του χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Ευτυχώς παρατήρησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα κράτη-μέλη, παρόλο που ισχυρίζονται θέλουν να επιλύσουν την κρίση με λύσει ευρωπαϊκέ, χρησιμοποιούν όλες τις δυνατές ρήτρες διασφάλισης ώστε αυτή η εποπτεία να μην μπορεί να γίνεται χωρίς διακυβερνητικές συμφωνίες. Δουλέψαμε όλοι καλά μαζί, αλλά δώσουμε στον καθένα αυτό που του ανήκει ως ε, εισηγήτρια για το συστημικό κίνδυνο, ο Μισελ Μπαρνιέ μιλάει πολύ για ραντάρ και πύργους ελέγχου, αλλά υπάρχει και ένας πιλότος αεροπλάνο. Αυτός είναι ο πρόεδρος της BCE, ε, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και αυτό θέλουμε να εξακολουθεί να ισχύει. Καλό λοιπόν όλους να συνεχίσουν τον αγώνα σε ό,τι αφορά την άμεση υποπτία των πανευρωπαϊκών οργανισμών και οντοτήτων. Στους Στα τομεακά κείμενα και τα τέσσερι βασικές ομάδες του Κοινοβουλίου το έχουν αναλάβει αυτό να δώσουν εξουσίες σε ό,τι αφορά του οίκους αξιολόγησης και ε, περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει συνέχεια στο θέμα αλλά και στον οργανισμό συμψηφισμών και στις διασυνοριακούς ομίλους. Ο αγώνας είναι ξεκάθαρος. Ή θα έχουμε μια εσωτερική αγορά με ευρωπαϊκή εποπτεία και ρύθμιση ή θα αρκουκεστούμε σε ένα συντονισμό πασαλήματα δηλαδή μεταξύ των διαφόρων ε, ε, κυρίαρχων χωρών. Ευχαριστώ την κυρία Μπουλάρ που χρησιμοποίησε βελγική ορολογία και θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο για ε, δυόμιση λεπτά. Ευχαριστώ. Καταρχάς, ήταν σημαντική στιγμή αυτή για την Ευρώπη. Από ό,τι φαίνεται συμφωνούμε πλέον για την εποπτεία. Πετύχαμε πολλά από κοινού και ευχαριστώ πολύ τη Βελγική Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κύριε Μπαρνιέ και τους συναδέλφους των διαφόρων πολιτικών ομάδων, τους συζητητές. Γιατί κάναμε πραγματικά ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Και αποδείχτηκαν ε, ότι είχαν άδικο εκείνοι που διαφωνούσαν με τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. Είμαστε όντως σε καλό δρόμο. Ε, αυτό ήταν το ένα που ήθελα να πω. Ένα δεύτερο. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα την παρακολούθηση των προπολογισμών των κρατών μελών. Αποφάσισε σημαντικά πράγματα το ΕΚΟΦΗΝ και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προτάσεις. Τώρα περιμένουμε και άλλες προτάσεις μακροοικονομικού συντονισμού. Επιγόντω χρειάζεται αυτό λόγω και της κρίσης. Τώρα επιτρέψτε μου να πω κάτι άλλο για το φόρο των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είδαμε κακοφωνία. Από τη μια ο κύριος Μπαρνιέ και ο κύριος Μπαρόσο καλά κάνουν και τους ευχαριστούμε και υποστηρίζουν. Ο κύριος Σεμετά όμως την απορρίπτει. Και παρακαλώ, συντονιστείτε, λειτουργήστε και εκεί συλλογικά με μία φωνή δεν μπορεί ο κύριος σε μετά να βγαίνει και να λέει τέτοια πράγματα και να κάνει και εκθέσεις όπου βγάζει διάφορα πορίσματα τα οποία έχουν καταρριφθεί επιστημονικά. Μπορεί να διαβάσει κανείς στην τη μελέτη που έχει αναθέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία καταρρύπτει τα επιχειρήματα του κυρίου Σιμετά. Και διαρωτώ με γιατί απουσιάζει σήμερα. Επανειλημμένα έχει ασκηθεί κριτική εις βάρος του. Τώρα γιατί δεν ήρθε να αντιμετωπίσει τη συζήτηση ο κύριος Σεμετά. Και κάτι άλλο. Είπαμε ότι θα καθίσει να τα ξανασκεφτεί και να τα ξανακοιτάξει αυτά. Ωραία. Και αυτό θα οδηγήσει σε καμία πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα αναλάβετε καμιά πρωτοβουλία ή μήπω θα ξαναβγεί μια μελέτη για ένα έγγραφο και μόνο. Γιατί δεν αρκεί αυτό. Και κάτι άλλο που δεν αρκεί είναι η απόφαση του Συμβουλίου που το παραπέμπει αυτό στο G20 όπου θα προεδρεύει η Γαλλία. Και αυτό δεν μας αρκεί. Και ε, οι κεντρικές χώρες που το αρνήθηκαν αυτό, η Μεγάλη Βρετανία και η Σουηδία και η Ισπανία. Το ξέραμε για τους δύο πρώτους, αλλά η Ισπανία είναι Eurogroup και ε, κυβερνάνε οι σοσιαλδημοκράτες εκεί. Δεν μπορείτε να συντονίσετε λίγο τη θέση σας με αυτά που λέτε εδώ και αυτά που λέει η Ισπανική κυβέρνηση στο Συμβούλιο. Και ένα τελευταίο. Εδώ στο Κοινοβούλιο θα περίμενα μεγαλύτερη σαφήνεια και θα επιθυμούσα και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ποια είναι επιτέλους η θέση σας. Ε, εκφράσατε μεγάλες επικρίσεις για την ε, επιβολή φόρου στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Πολλοί όμως από την ομάδα σας είναι υπέρ. Δεν ξέρω κυρία Βόρτμαν Κόλλαν ε, εκπροσωπείτε την πλειοψηφία των συναδέλφων σας. Αλλιώς οι πολίτες θα μας αντιμετωπίζουν με κινησμό. Γιατί έχουμε πακέτα λιτότητας και εξοικονόμησης, αλλά στις τράπεζες τις αφήνουμε να αλωνίζουν. Η κυρία Σούνιμπερ έχει τώρα το λόγο, παρακαλώ. Για 1,5 λεπτό. Thank you. I'd like to... Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τη Βελγική Προεδρία για την διαπραγμάτευση και τον Επίτροπο Μπαρνιέ γιατί βρήκε λύσεις για την εποπτεία. Αλλά πολλά θέματα δεν λύθηκαν χτες στο ΕΚΟΦΗΝ. Στο Κοινοβούλιο ζήτησαν να διενεργηθεί ε, έρευνα αντικτύπου και είδαμε ότι το ΕΚΟΦΗΝ ακριβώς αυτό έκανε χωρίς να λάβει υπόψη τα πολιτικά δεδομένα και να νομοθετήσει. Λάβαμε υπόψη στατιστικά δεδομένα, καλύτερη ρύθμιση, έμπρακτα. Όμως, όταν ένας ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας είπε ότι θα συλλέξει το 70% από τα έσοδα από αυτή τη φορολόγηση, είναι γελίο να ζητήσετε αυτό να επιβληθεί σε ε, ε, ευρωπαϊκό επίπεδο. Το, οι, οι ενδιάμεσοι μεσάζοντες δεν πρέπει να καταβάλουν το ε, αντίκτυπο, το αντίτιμο, με συγχωρείτε, για αυτή τη φορολόγηση. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τους περιορισμούς αυτού του απλουστευμένου FTT και δεν θα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη αυτό τον φόρο συναλλαγής ε, ο οποίος θα επιβληθεί σε όλους. Αντί να υπάρξει εκτροχιασμός μέσα στα πλαίσια αυτής της συνολικής, του συνολικού φόρου συναλλαγής θα πρέπει να αδράξουμε αυτή την ευκαιρία για να αντιμετωπίσουμε τα αδύναμα οικονομικά μας και τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν το θέμα ε, σε κρατικό επίπεδο. Ο κύριος Πόρτας για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ. Το ΕΚΟΦΗΝ αποφάσισε να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό εξάμεινο και να λάβει υπόψη μία συνοχή που θα πρέπει να ισχύσει σε δημοσιονομικό επίπεδο. Λάβατε υπόψη τις ε, δημοκρατικές αρχές. Δέχομαι μέτρα αντιμετώπισης του ελλείμματος, αλλά να δημιουργείται και απασχόληση. Δέχομαι βελτιώσεις των εθνικών προϋπολογισμών, αλλά δεν πρέπει τα μέτρα να είναι ιδιαίτερα αρνητικά δημοσιονομικά. Δεν, μπορεί, δεν μπορούν οι Βρυξέλλες να αποφασίσουν πώς θα εκπληρώσουν τα κράτη-μέλη αυτούς τους όρους. Διότι αυτό σημαίνει ότι αποκηρύσουμε την εθνική μας κυριαρχία. Δηλαδή το ΕΚΟΦΗΝ στην ουσία ορίζει κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να ορίζουν κάθε εθνικό προϋπολογισμό. Μας είπε η Προεδρία, μα δεν θα πούμε σε λεπτομέρειες. Δέχομαι τη μεγαλοθυμία του, όμως οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές θα οριστούν από τις 27 κυβερνήσεις και η Γερμανία πάντα θα λέει στους Έλληνες τι πρέπει να κάνουν. Αλλά το αντίθετο δεν μπορεί ποτέ να συμβεί. Η ε, εθνική ε, οι βουλευτές του Εθνικού Κοινοβουλίου δεν μπορούν να απαρνηθούν την εθνική τους κυριαρχία και την ελευθερία επιλογών. Ευχαριστούμε και το λόγο έχει ο Hans Peter Μάρτιν για ένα μισή λεπτό. Κύριε Επίτροπε, στα γαλλικά και τώρα στα γερμανικά, να σας κάνω μια φιλοφρόνηση. Φαίνεται ότι επιθυμείτε ε, να προχωρήσετε. Τίστε το ερώτημα όμως σας επιτρέπετε να επιθυμείτε. Έχετε μεγάλη προσήλωση στο καθήκον σας. Αλλά παρακαλούσα να δείχνετε την ίδια φάνεια και προς τους πολίτες. Τη διαφάνεια και τη σαφήνεια και να εξηγήσετε γιατί αποτυχάνετε ακόμα και αν έχετε καλή βούληση. Και στις τέσσερις πυλώνες και τα βασικά ζητήματα είναι περιορισμένη η πρόοδος που έχει γίνει. Χρειάζεται διαλεύκανση αυτού. Η χρηματοπιστωτική εποπτεία σε ουσιαστικού τομεί στι Ηνωμένε Πολιτείε είναι και πιο κρίσιμη και πιο αυστηρή σε σχέση με αυτά που προσπαθείτε τώρα να στήσετε. Χρειαζόμαστε λοιπόν σαφεί απαντήσει και στο μέλλον. Τι θα κάνετε με τις ε, γκρίζες ζώνες και τις ε, σκιώδεις τράπεζες και τι θα γίνει με το ίδιο κεφάλαιο. Τι θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει. Είναι πάρα πολύ μεγάλες οι λεπτομέρειες και πού θα οδηγηθούμε. Να μην έχουμε ξανά τέτοια φαινόμενα, τέτοια κράση. Και εγώ που είμαι από μια μικρή χώρα, θέλω να ρωτήσω τι μπορεί κανείς να κάνει για να περιοριστεί αυτή η προβληματική το too big to fail. Έχουμε μια τράπεζα, ας πούμε, που ε, ε, μπορεί μια τράπεζα να κάνει το χρέος της Αυστρίας να φτάσει σε επίπεδα τύπου Ελλάδας. Πώς θα αποτρέψετε εσείς η Αυστρία να είναι δεύτερη Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, κύριε Μάρτιν. Παίρνουμε τώρα τους επόμενους εγγεγραμμένους ομιλητές, ξεκινώντα από τον κύριο Γκόζδες. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να συγχαρώ κι εγώ για τα καλά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σε θέματα εποπτείας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασφαλώς συνέβαλε σε αυτό και το Δεκέμβριο μοναδικό γεγονός και νέο γεγονός είχαμε μια δήλωση των τεστάρων συντονιστών των κυριωτέρων ομάδων οι οποίοι έλεγαν ότι χρειάζεται αυτή την εποπτεία περισσότερη Ευρώπη. Ο δυναμισμός σας κύριε Υπουργέ επέτρεψε να καταλήξουμε σε μια ικανοποιητική λύση. Η Επιτροπή εργάστηκε και εκείνη πολύ και χαιρετίζω το πρόγραμμα που μας ανακοίνωσε ο Επίτροπος Μπερνιέ σε ό,τι αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Ευτυχώς που επετεύχθη αυτή η συμφωνία, διότι τελικά σε θέματα χρηματοπιστωτικά αυτό που έχει σημασία είναι η αξιοπιστία της Ευρώπης. Αξιοπιστία έναντι των πολιτών μας, οι οποίοι μα ρωτούν από τότε που προέκυψε η κρίση τι κάνει η Ευρώπη, ποια είναι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα στα οποία καταλήξατε. Λέμε ότι έχουμε συνεδριάσει, συναντήσει, τριμερίσει επαφέ, αλλά αυτά που θέλουν αποτελέσματα και η αξιοπιστία τη Ευρώπη έναντι των διεθνών εταίρων μα και των Ηνωμένων Πολιτειών ειδικότερα. Πρόσφατα είχα επαφέ με του, του χρηματοπιστωτικού τομέα των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτό που του ανησυχεί και που φοβούνται κάπω στην Ευρώπη είναι η εντύπωση, αυτή η εντύπωση της ε, δικαστικής ε, νομικής ανασφάλειας. Αλλάζουν τα συστήματα, ε, έχουμε διάφορες ρήτρε, sunset clause, χωρίς όμως κάτι το πολύ συγκεκριμένο. Πρέπει να καταλήξουμε σε ένα σύστημα το οποίο θα είναι οριστικό, χωρίς να δώσουμε την εντύπωση ότι μετά από δύο-τρία χρόνια κάτι θα αλλάξει. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα λοιπόν να ε, ζητήσω το εξή. Σήμερα το απόγευμα θα γίνει μια πολύ σημαντική τριμερή συνάντηση με τον κύριο Μπαρνιέ και άλλου συναδέλφου για τα εναλλακτικά ταμεία. Πρέπει, είναι απαραίτητο να βρούμε γρήγορα μία λύση. Ξέρω πόσο πολύ έχει δεσμευθεί η Βελική Προεδρία και εσείς προσωπικά. Τις επόμενε εβδομάδε πρέπει να καταλήξουμε σε μία συμφωνία ώστε την επόμενη φορά που θα λογοδοτήσετε για το εργασίε του ΕΚΟΦΗΝ να μπορέσετε να μας πείτε έχουμε βρει, έχουμε βρει μια λύση για το θέμα των εναλλακτικών ταμείων. Νομίζω ότι θα κάνετε ό,τι χρειάζεται για να βρεθεί η πιο σωστή λύση. Ευχαριστώ. Η κυρία τώρα το λόγο. Για λεπτό Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, οι χθεσινέ αποφάσει του ΕΚΟΦΗΝ σε συνδυασμό βεβαίω με τη συμφωνία για, για ένα αποτελεσματικό σύστημα χρηματοπιστωτική εποπτείας αποτελούν ουσιαστικά βήματα προ την κατεύθυνση τη νέα οικονομική διακυβέρνηση που οραματιζόμαστε όμως η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι ευρύτερη δεν μπορεί και δεν πρέπει να σταματά στην αυστηροποίηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της εποπτείας. η πρόκληση είναι η διαμόρφωση ενός νέου οικονομικού μοντέλου που θα δίνει απαντήσεις στο αίτημα των ευρωπαίων πολιτών για πλήρη απασχόληση και για δίκαιη ανάπτυξη. χρειάζεται λοιπόν να διασφαλίσουμε μια ισορροπία ανάμεσα στη δημοσιονομική πειθαρχία και την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για βιώσιμη ανάπτυξη και για πλήρη απασχόληση με επενδύσει, δημόσιες και ιδιωτικές. χρειάζεται ασφαλώ να αντιμετωπίσουμε τις μακροοικονομικές ισορροπίες και το χάσμα ανταγωνιστικότητας μεταξύ των κρατών μελών που οδηγεί αναπόφευκτα σε οικονομικές και κοινωνικέ ανισότητε. πάνω απ' όλα όμω, χρειαζόμαστε ένα μοντέλο δικαιότερης κατανομής του κόστους της ανάκαμψης και φορολογικής δικαιοσύνης και εδώ η φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών μπορεί να παίξει ένα ρόλο καταλυτικό. η ευρώπη μπορεί και πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο θέμα αυτό το έκανε με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και δεσμεύτηκε μονομερώς μπορεί και πρέπει να ηγηθεί της προσπάθειας να προωθηθούν αντίστοιχες ρυθμίσεις στο διεθνές επίπεδο. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Ποδηματά. Ο Ρόντ. Ένα λεπτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να υποστηρίξω και να συγχαρώ την Επιτροπή και το Συμβούλιο για τις ε, προσπάθειές τους σε ό,τι αφορά το θέμα της φορολόγησης εμείς θέλουμε να εξασφαλιστεί ένας ε, συντονισμός και σταθερότητα. Όταν μιλάμε όμως για τέτοια φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, μιλάμε για ένα πολύ πιο σύνθετο φόρο. Θα χρειαστεί να είναι σφαιρικός, ε, να καλύπτει όλες ε, και η φορολόγηση όλων των συναλλαγών μπορεί να, μπορεί να μην είναι κάτι το εφικτό και μπορεί να αυξήσει και την μεταβλητότητα και την αστάθεια των αγορών. Εάν ο σκοπός είναι να συγκεντρώσουμε χρήματα για παγκόσμια προγράμματα, ποιος θα είναι υπεύθυνος για την κατανομή, για τον επιμερισμό αυτών των χρημάτων. Και πότε θα ξέρουμε ότι τα χρήματα έχουν πλέον, είναι πλέον επαρκή. Ποιο θα αναλάβει το συντονισμό όλη αυτή τη διαδικασία, τα κράτη ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση μακριά από του πολίτε τη, πώ θα αποτρέψουμε την συνεχή αύξηση τη φορολόγηση. Γιατί στον πραγματικό κόσμο το αρκετό δεν είναι ποτέ αρκετό όταν μιλάμε για τις ανάγκες, ανάγκες των πολιτικών για περισσότερα χρήματα. Ευχαριστώ κύριε Ρόντ. Ο κύριος Έπινγκ τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Ρέντερς. Ελπίζω να είστε καλά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με το φόρο των τραπεζών, αλλά διαρωτώ με πώς μπορεί ε, να προχωρήσει. Ε, όταν είσαι σε ένα λεωφορείο, όλοι είναι υπέρ του λεωφορείου, αλλά θέλουν να το στρέψουν σε άλλη κατεύθυνση. Για το φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών είναι κακή ιδέα. Δεν μπορούμε να έχουμε ε, ευρωπαϊκό φόρο Τόμπιν και δεν μπορούμε να μιλάμε για φόρο Τόμπιν γιατί ο ίδιος ο Τόμπιν πλέον είναι κατά του φόρου Τόμπιν. Οπότε τι θα γίνει, θα μας φύγουν κεφάλαια, δεν θα έχουμε έσοδα και πού είναι ήδη οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα γίνει μεγάλη φασαρία. Κύριε Ρέντερς, σας δίνω καλόπιστη ε, συμβολή. Σταματήστε το, βάλτε στο ψυγείο για να μην μπω στο καταψύκτη αυτό το θέμα. Και ο κύριο Σούλτς που δεν με ακούει είχε πει ε, ε, χτες ότι θέλει να αναγκάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία για το φόρο ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και θα κινητοποιήσει και τον κόσμο. Μην το κάνετε, γιατί ο πολίτης θα το πληρώσει. Και εμεί θα ξεκινήσουμε μια πρωτοβουλία πολιτών προς την κατεύθυνση αυτή, αντίθετη δηλαδή. Ο κύριος Κάρας, για δύο λεπτά. Κύριε Επίτροπε, κύριε Προεδρεύον του Συμβουλίου, κυρία Πρόεδρε, έχω πέντε σημεία να σας αναφέρω. Πρώτον, θα πρέπει να πω ότι λυπάμαι που μια τόσο σημαντική συνεδρίαση του ΕΚΟΦΗΝ όπως ήταν χτεσινή διεξαγόταν παράλληλα με την ομιλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ περιμένω καλύτερο συντονισμό των εργασιών μας. Αν θέλουμε να πηγαίνουμε ε, όλοι προς την ίδια κατεύθυνση θα πρέπει από κοινού ε, να ε, προχωρούμε, να συντονιζόμαστε, να ακούμε ένα τον άλλον και να συνομιλούμε. Ήταν μια άχρηστη παράλληλη συνεδρίαση που μας αποδυνάμωσε. Δεύτερον, ευχαριστώ πολύ την Προεδρία και το ε, Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εποπτεία. Αν δεν υπήρχε απόφαση του Κοινοβουλίου τον Ιούλιο, δεν επρόκειτο να είχαμε καταλήξει πουθενά. Θα είχαμε χάσει τις προθεσμίες αν δεν είχε αποφασίσει ε, το ε, κοινοβούλιο τον Ιούλιο, ούτε ο πρόεδρος τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήταν τώρα πλέον πρόεδρος τη Εποπτείας. Δείξαμε τα δόντια μας, σκληρίναμε τη στάση μας και πραγματικά αυτό βοήθησε και μας υποστήριξε και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Σημείο τρίτον. Ναι, στον εξευρωπαϊσμό της συζήτηση ε, για τον προπολογισμό των κρατών αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι το δεύτερο σκέλος της νομισματικής ένωσης, η οικονομική δηλαδή, θα πρέπει να είναι οικονομική και η κοινωνική ένωση και αυτό θα γίνει με πολιτικές ε, ε, προϋπολογισμού και φορολογικές πολιτικές και να είναι ευρωπαϊκές, όχι ε, απλό συντονισμό. Τέταρτο, ευρωπαϊκή στόχη και δημιουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου και πέμπτο για το φόρο των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, σιγά σιγά ε, θα πρέπει να το προωθούμε αυτό το θέμα. Κύριε ε, Προεδρεύον, είπατε ότι ήταν η πρώτη σοβαρή συζήτηση. Εδώ και ένα χρόνο το συζητάμε εμείς. Κάνουμε ερωτήσει, ψηφίσματα επιψηφισμάτων. Και εσείς Παίζετε την κολοκυθιά. Πότε το G20, πότε τα κρατημέλη, πότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απαντήστε επιτέλους. Ε, ποιος, ε, ε, ποιο είναι το ποσοστό, ποιος είναι ο συντελεστής, ποια είναι η βάση φορολογική, ποιος θα πάρει τα χρήματα και τι θα τα κάνει. Κάντε ένα σχέδιο, εν περιπτώσει, για να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ, κυρία Φεραίρα. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συντονιστούν οι προσπάθειές μας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που αποτέλεσε αντικείμενο ανάλυσης από το χτεσινό ΕΚΟΦΗΝ, αλλά είναι μόνο ένα μέρος της πραγματικότητας. Θα πρέπει η ανάπτυξη και η απασχόληση να αποτελέσουν προτεραιότητες μαζί με το Σύμφωνο Σταθερότητας. Θα πρέπει να δημιουργηθούν ε, ε, νέες θέσεις απασχόλησης και να αντιμετωπίσουμε και το ε, κυρίαρχο χρέος. Θα πρέπει να προωθήσουμε αυτή την εργασία και δεν θα πρέπει να θα στα πλαίσια των κυρώσεων. Ο κύριος Μπαρνιέ θα μπορέσει να μας βοηθήσει με την πολύχρονη πείρα του. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω στα πλαίσια, για την εργασία στα πλαίσια της ε, χρηματοπιστωτικής εποπτείας ο Επίτροπος Μπαρνιέ μαζί με το Κοινοβούλιο και τη Βελγική Προεδρία φτάσανε σε μια πολύ καλή συμφωνία που μας τιμά και που προασπίζει τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Ελπίζω να ακολουθήσουμε την ίδια μεθοδολογία και στο μέλλον. Έπειτα, στη συνέχεια, θα ήθελα να πω προς τον Επίτροπο ότι ως προς το σύστημα εξυγίανσης και αντιμετώπισης συστημικού κινδύνου θα μπορέσετε να αποτιμήσετε την ευρωπαϊκή διάσταση του φαινομένου. Τέλος, θα πρέπει να ξαναδούμε την ατζέντα μας για τους G20, ιδιαίτερα αν δεν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την απάτη και την φορολογική ε, αποφυγή. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεισφέρουν οι τράπεζες και να καταβάλουν εκείνες το αντίτιμο των πράξεών τους. Έληξε ο χρόνος σας. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Φόρντ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Χαιρετίζω τη συμφωνία και είμαι βέβαιη ότι ήταν δύσκολο να καταλήξουν οι συνάδελφοι στη συμφωνία. Χρειάστηκε να βρεθεί μια λεπτή ισορροπία για την προστασία των αγορών Αφενό και την διατήρηση των ε, αρμοδιοτήτων των κυβερνήσεων. Το είπε, όπω είπε πολύ σωστά ο Επίτροπος, είναι το πρώτο στάδιο και προσβλέπω στη συνεργασία με τους Επιτρόπους ώστε με τα, στα επόμενα στάδια να μην διαταραχθεί αυτή η λεπτή ισορροπία. Τα κράτη-μέλη να, δεν μπορούν να συμφωνούν διεθνώς για πρότυπα και να μην είναι σε θέση να τα εφαρμόσουν σε εθνικό επίπεδο. Όλοι πρέπει να τηρούμε τα διεθνή πρότυπα. Στη συζήτηση πολλοί συνάδελφοι είπαν ότι είναι σημαντικό ο αρχηγός, ο επικεφαλής του Οργανισμού Διεθνών Λογιστικών Προτύπων να συνεργάζεται στενά με την Κεντρική Τράπεζα. Ειδοποίησε χθες το Συμβούλιο για τους κινδύνους που θα μπορούσε να έχει για την Ευρώπη η επιβολή αυτού του φόρου πάνω στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Είναι λοιπόν σημαντικό να, ε, ε, να ακούμε αυτά που έχουν να μας πούν ορισμένοι. Κυρία Οκονή τώρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως είπαν και οι άλλοι συνάδελφοι και ο Ζων Γκοζές πριν από λίγο ή χθε στη διάρκεια της συζήτησης για την κατάσταση της Ένωσης χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Περισσότερη Ευρώπη για να δημιουργήσουμε ανάπτυξη και θέσει εργασία για να ρυθμίζονται και να σταθεροποιούνται αγορές και να μειώνονται οι ανισότητες. Όπω τόνισε και ο πρόεδρο τη ομάδα μου, ο Ζωζεφ Ντόλ, με τον οποίο συμφωνώ απόλυτα. Τα κράτη-μέλη ελπίζω ότι κατάλαβαν επιτέλου, ότι στον δημοσιονομικό και χρηματοοικονομικό τομέα πρέπει να είμαστε τολμηροί και υπεύθυνοι. Οι προστατευτικές τα προστατευτικά αντανακλαστικά δεν ωφελούν κανένα. Χρειαζόμαστε περισσότερη χρηματοοικονομική εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η συμφωνία με το Συμβούλιο για τη, τη δέσμη ε, της χρηματοοικονομικής εποπτείας που θα ψηφίσουμε στην επόμενη Ολομέλεια είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Αλλά πέρα από την εποπτεία του συστήματος, αυτό που χρειάζεται είναι ουσιαστικό συντονισμό των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών μας. Πρέπει να καταλήξουμε σε έναν δημοσιονομικό και οικονομικό ομοσπονδιακό σύστημα. Όταν είμαστε ενωμένοι για μια νομισματική πολιτική αλλά αυτόνομη σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές μας δεν καταλήγουμε σε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Το ευρωπαϊκό, το το ευρωπαϊκό εξάμεινο που υποχρεώνει τις χώρες να υποβάλουν τον προπολογισμό τους κάθε χρόνο πριν από το καλοκαίρι. Γι' αυτό θα, η πρακτική θα καθιερώσει και θα υποδείξει ποιο είναι το σύστημα που μπορεί να εφαρμοστεί πολύ καλύτερα από ότι τα κείμενα. Στον τομέα της οικονομικής και βιομηχανικής πολιτικής αλλά και στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής λυπάμαι που τα Εθνικά Κοινοβούλια αλλά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμμετέχουν πλήρως σε αυτή τη διαδικασία συντονισμού. Κύριε Υπουργέ, ως, ως εκπρόσωπο του Συμβουλίου απευθύνομαι ειδικότερα σε εσά ως αρμόδια αρχή για τον προπολογισμό τα ευρωπαϊκά τα κοινοβούλια πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην χάραξη μιας ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής γιατί εξαρτάται από αυτό η αξιοπιστία και η νομιμότητα. Θα σας διακόψω τώρα και θα δώσω το λόγο στον κύριο Σάντσες Πρεζέντο για 1,5 λεπτό και τον παρακαλώ να τηρήσει το χρόνο του. Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Προεδρία για την ομοφωνία που επέτυχε το Συμβούλιο και το συμβιβασμό ως προς το πακέτο εποπτείας. Ε, ε, εργαστήκαμε ήδη από την Ισπανική Προεδρία και με τη Βελγική και φτάσαμε σε έναν φιλόδοξο συμβιβασμό που θέτει τα θεμέλια της οικονομικής μεταρρύθμισης και ολοκληρώνει την, και φτάνει στην ολοκλήρωση της Ευρώπης. Μιλήσαμε για το ευρωπαϊκό εξάμεινο του επόμενου έτους, αλλά είναι δύσκολο να ορίσουμε ένα χρονοδιάγραμμα ενεργειών και να προσδώσουμε σε αυτές ε, καθαρά ε, κοινοβουλευτικό χαρακτήρα. Πρόκειται για θέμα οικονομικής διακυβέρνησης. Θα πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα της οικονομικής ανάπτυξης με βάση την ε, και την κοινωνική συνιστόσα θα πρέπει να προλαμβάνουμε και να επιλύουμε τις κρίσεις, να ορίσουμε ένα εύρωστο σύστημα έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους και τους κινδύνους δεοντολογίας και να αποφύγουμε στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά. Θα πρέπει να συντονιστούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και στους G. 20. Και ως προς την φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών αναμένουμε την ε, πρόταση της Επιτροπής έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τους κλειδονισμούς και την κρίση των δημοσίων οικονομικών και να προσλάβουμε νέους πόρους για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα πλαίσια της πλήρωσης των στόχων της χιλιετίας. Το λόγο έχει ο κύριος Σκίνερ για μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κύριε Ρέιντερς, Επίτροπε Μπαρνιέ, σας ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη του πακέτου εποπτείες και φαινόταν σαν να ψάχνουμε ψήλου στάχυρα στην ουσία. Ελπίζω να μπορέσουμε να είμαστε πιο παραγωγικοί μέσα στα πλαίσια των μέτρων εφαρμογής του πλαισίου. Υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία, αλλά και πολλά αρνητικά που υπογραμμίστηκαν. Όμως, συμφωνώ με την πρόοδο που έχει επιτελεστεί η Ευρώπη όμως δεν είναι μόνο η Ευρωζώνη. Πρέπει να, έχουμε, ε, να βρούμε τρόπο αποδοτικότητας στο, στην εφαρμογή των κανονισμών. Δεν είμαστε φυγόδικοι. Έτσι αισθάνονται ορισμένα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν σύνολο και να δούμε και τη διεθνή μας ατζέντα θα πρέπει να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο για να φτάσουμε σε παγκόσμιους στόχους. Αν πιστεύουμε ότι με τα ευρωπαϊκά πρότυπα αυτό αργεί, τότε κάνουμε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Γι' αυτό καλωσορίζω τα σχόλια του Επιτρόπου Μπαρνιέ για, το, για παράλληλη, μια παράλληλη πορεία ως προς την εποπτεία και θα θέλαμε να δούμε το περιεχόμενο αυτής της μελέτης σας, κύριε Επίτροπε. Θα ήταν πολύ χρήσιμο. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο. Πώς θα κινηθούμε στο μέλλον. Έχουμε προβλήματα ενώπιον μας που δεν μπορούμε να επιλύσουμε μόνοι μας. Ευχαριστούμε κύριε Σκίνερ. Ο κύριος Βαν Κόκ έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, το Συμβούλιο Εκοφίνε χτες ενέκρινε την αρχή του λεγόμενου ε, Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ως φεντεραλιστής δεν μπορώ παρά να χαροποιούμε από μια τέτοια πρόοδο. Αλλά ο συντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών είναι ε, ε, με ένα θέμα, αλλά το περιεχόμενο τους και πώς θα ορίζεται είναι μια άλλη υπόθεση. Και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης εδώ είναι μεγάλο σφάλμα έχω επιβληθεί με ένα δογματισμό μια κούρα λιτότητα σε όλη την Ευρώπη και δίνει τα αποτελέσματα. Η Ισπανία και η Ιρλανδία βαθίζονται όλο περισσότερο στις δυσκολίες. Και τέλη ε, Αυγούστου μια μελέτη Market έδειξε ότι ε, η ε, ανάπτυξη στην Ευρώπη και στη Γερμανία σε λίγο αποτελματώνεται. Κατασταλτικά μέτρα διαφαίνονται στο άτυπο ΕΚΟΦΗΝ που ακολουθεί και είναι ακόμα πιο σοβαρά αυτό. Να επιβάλλονται κυρώσει σε χώρε που ήδη αντιμετωπίζουν δημοσιονομικό πρόβλημα είναι ανεύθυνο. Πηγαίνουμε κατευθείαν σε σύγκρουση με το θέμα των πόσο συμβάλλουν στον κοινοτικό προϋπολογισμό ε, τα κράτη-μέλη. Χθε βγήκαν στον δρόμο 2,5 εκατομμύρια Γάλλοι. Θα πρέπει να διατηρηθούν οι κοινωνικές αντιστάσεις και να υπάρξει να διασφαλιστεί κοινωνική ειρήνη που χρειάζεται για να ανακάμψει η οικονομία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι πυρομανή στη στάση της. Υπάρχει ευρωσκεπτικισμός όλο και μεγαλύτερος στη στάξη των πολιτών. Στο όνομα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και στην υπηρεσία των πολιτών που γι' αυτά, αυτούς γίνονται όλα αυτά, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι οικονομική ανοησία ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας, αλλά ταυτόχρονα και μέγα πολιτικό σφάλμα. Ευχαριστώ πολύ και τώρα ακολουθεί η διαδικασία Catch Δηλαδή, ε, έχουν ζητήσει το λόγο διάφοροι συνάδελφοι και θα τους το δώσω. κύριος Νίτρας για ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ. Με ιδιαίτερη χαρά Χαιρετίζω την συμβιβαστική λύση για την χρηματοπιστωτική εποπτεία. Πράγματι, οι ευρωπαϊκές αγορές απαιτούσαν, ζητούσαν έναν τέτοιο μηχανισμό. Και αυτό που με ικανοποιεί αυτή την απόφαση είναι ο ρόλος που θα αναλάβει, που θα παίξει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι η εμπειρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζα θα μας επιτρέψει να ατενίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό εξάμεινο είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Έτσι, με ουσιαστικό τρόπο θα συντονίζουμε την οικονομική πολιτική αλλά και τις ευρωπαϊκές δαπάνες. Και κάτι πολύ πιο σημαντικό, ε, το σύστημα του reporting, της ε, υποβολής εκθέσεων. Τα κράτη-μέλη που λαμβάνουν αποφάσεις δεσμεύονται με αυτό το σύστημα να σέβονται το δημοσιονομικό σύστημα. Πρέπει να σας διακόψω κύριο Σκυτάς τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Πιστεύω ότι το σύμφωνο σταθερότητας θα πρέπει να αναθεωρηθεί, καθώς και το οικονομικό μας μοντέλο. Έχει μία ιδειτερότητα και γι' αυτό θα πρέπει να τύχει υποστήριξης. Μιλήσαμε για ε, μία ατμομηχανή οικονομικής ανάπτυξης, η οποία όμως απέτυχε στις προσδοκίες. 10% Ευρωπαίοι δεν έχουν θέση εργασίας και βλέπουμε ότι υπάρχει ύφεση παντού. Επίσης υπάρχει μεγάλο έλλειμμα το οποίο ε, έθεσε στην επιφάνεια, έφερε στην επιφάνεια οικονομική κρίση. Γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, διότι πιστεύω ότι το κοινό νόμισμα και η αγορά θα μας βοηθήσει. Χαιρετίζω τις αποφάσεις του ΕΚΟΦΗΝ και ιδιαίτερα την μακροοικονομική εποπτεία, καθώς και την Επιτροπή Εποπτείας και Αντιμετώπισης Συστημικού Κινδύνου. Και επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να εποπτεύσουμε τα ευρωπαϊκά θέματα μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ε, εξαμήνου. Η κυρία Φιγκεϊρέδο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι απαράδεκτες οι χτεσινές αποφάσεις του Συμβουλίου ΕΠΟΦΗΝ. Οι κερδοσκόποι παραμένουν με ανοιχτά τα χέρια και πλήρως ελεύθεροι να δράσουν όπως θέλουν. Η φορολόγηση δεν λύνει το πρόβλημα, διότι όλες οι πλούσιες χώρες χρησιμοποιούν ως πρόφαση την κρίση για να κερδοσκοπήσουν. Είμαστε μαριονέτες γιατί μιλάμε για φορολόγηση όπως την ορίζει το Ευρωπαϊκό Διευθυντήριο, σαν να μην έφτανε το σύμφωνο σταθερότητας και τα παράλογα κριτήριά του. Πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις συνθήκες που δεν ε, ορίζουν την καταπάτηση της εθνικής κυριαρχίας, που είναι νευραλγική σημασίας. Και χτες προωθήθηκαν τα συμφέροντα των μεγάλων οικονομικών μπλοκ και αυτό θα έχει ολέθριες συνέπειες στα οικονομικά της Ευρώπης. Πιστεύω ότι η μάχη των εργαζομένων θα εντατικοποιηθεί. Τέλος, η κυρία Γιάν Κοσάρη έχει το λόγο για ένα λεπτό επίσης. Ευχαριστώ ε, πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο στη διαδικασία αυτή. Πριν από μερικά χρόνια επικράτησε ο νεοφιλελευθερισμός και ε, το δόγμα ήταν να μην ανακατεύεται η πολιτική στην αγορά, η αγορά θα τα ρυθμίσει από μόνη της. Τώρα έχουμε καταλάβει όμως ότι η πολιτική έχει ένα ρόλο να διαδραματίσει, να παίρνει αποφάσεις και να θέτει τα πλαίσια. Το είδαμε στην εποπτεία, το είδαμε και στα θέματα τα δημοσιονομικά ε, να υποβάλλονται ε, εκ των προτέρων οι προϋπολογισμοί και να είναι σωστά τα στατιστικά στοιχεία χωρίς μανούβρες και χειραγώγηση. Τώρα καταλαβαίνουμε τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό που είχε πει στο παρελθόν ο Σούμαν, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα τότε προχωρεί μέσα από κρίσεις. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του Catch the Eye και θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μπαρνιέ πρώτα, εξ ονόματος της Επιτροπής και μετά στον Προεδρεύμα του Συμβουλίου. Ευχαριστώ όλους σας και όλες σας για αυτά που είπατε για το συλλογικό αποτέλεσμα στο οποίο καταλήξαμε για την εποπτεία. Επανέρχομαι σε κάτι που είπε η κυρία Φεραίρα προηγουμένως, αναφερόμενη στους πολίτες, οι οποίοι πλήττονται από την κοινωνική, την οικονομική, τη χρηματοπιστωτική κρίση, την επιστημιστική, οικολογική κρίση οι πολίτες ε, μας εκλέγουν πρέπει να λογοδοτούμε σε αυτούς και να τους δείξουμε σαφώς ότι έχουμε αντλήσει διδάγματα από την κρίση. Όπως έγινε στην περίπτωση της εποπτείας πρέπει να, το, να εξηγήσουμε ε, ακριβώς. Ξεκινήσαμε με την έκδοση Μακάτι για το θέμα των αμοιβών. Θέμα με, παίρνοντας το, το ένα θέμα μετά το άλλο από αυτά που ταράζουν και προβληματίζουν τους πολίτες πρέπει να δείξουμε ότι ως Συμβούλιο, ως Κοινοβούλιο και ως Επιτροπή είμαστε σε θέση να δώσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο συγκεκριμένες απαντήσεις για τη φορολόγηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Έκανε πολύ σημαντικό έργο ε, ανάλυσης των διαφόρων κατευθύνσεων και των συνεπειών ε, από την ε, που θα υπάρξουν από την, μετά από την εφαρμογή αυτού του φόρου θα έλεγα στον κύριο Γκίγκολτ ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής έλαβε σαφώς θέση μιλώντας για μια ουσιαστική αλλά ίση και δίκαιη ε, κατανομή ο κύριος Καρά, κύριε δεν θα χρειαστεί να περιμένετε πολύ, ούτε, η συζήτηση αυτή συνεχίζεται. Δεν αρκεί να πιστεύουμε ότι έχουμε δίκιο εμείς και να το γνωρίζουμε. Πρέπει να πείσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες και τις 27 κυβερνήσεις και τις άλλες περιοχές του πλανήτη. Και αυτό θα απαιτήσει χρόνο και πολλή προσπάθεια. Όπως είπαν η κυρία Σουνίντεν, η κυρία Βανκόλ, η κυρία Φόρντ, αυτός ο φόρος για να είναι πραγματικά αποτελεσματικός πρέπει να εφαρμοστεί στην ευρύτερη δυνατή κλίμακα και για να γίνει αυτό πρέπει να πιστούν και οι άλλες περιοχές του κόσμου. Στον κύριο Σκίνερ θα ήθελα να πω ότι θα προετοιμάσουμε αυτό το συγκριτικό πίνακα αφού έγινε μεταξύ Αμερικανών και Ευρωπαίων, αφού γίνει μεταξύ Αμερικανών και Ευρωπαίων, πρέπει να στραφούμε και προς άλλες περιοχές του κόσμου. Την Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία, την Αφρική επίσης που έχει τη θέση και το ρόλο της και δέχεται πολλές συνέπειες. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν όλα τα στοιχεία στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Σκίνερ για τη διακυβέρνηση στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Ποδηματά και ο κύριος Μάρτιν δεν εφαρμόζουμε πάντοτε τις ίδιες μεθόδους, δεν έχουμε πάντα τους ίδιους νόμους, διότι οι οικονομίες μας είναι διαφορετικές μεταξύ τους. Ο κύριος Μάρτα αναφέρθηκε στην περίφημη στρατηγική του Βόλκερ. Εμείς έχουμε μια άλλη ανάλυση στην Ευρώπη. Ε, ε, ανάλογα με το μέγεθος και τις δραστηριότητες των τραπεζών αυτό που θέλουμε να υπάρχει εσωτερική και εξωτερική αποτελεσματική εποπτεία και διακυβέρνηση χωρίς να εμποδίσουμε, παρεμποδίσουμε την διαφορετικότητα και την ε, πολυμέρεια των δραστηριοτήτων τους. Επίσης, ο κύριος Νιτράς θύμισε τον σημαντικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της οποίας ο πρόεδρος θα είναι ο πρώτος πρόεδρος, ο οποίος θα δώσει αξιοπιστία στο Συμβούλιο Συστημικών Κινδύνων. Ο κύριος Καράς θύμισε ότι χάρη στην πρωτότυπη εξαιρετική απόφαση που πήρατε όλοι μαζί τον Ιούλιο να μεταφερθεί η ψηφοφορία σας για την πρώτη ανάγνωση στον φθινόπωρο, χάρη σε εσάς είχαμε το χρόνο να πείσουμε και το Συμβούλιο και να σημειώσουμε προόδους με το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους και θα κλείσω αναφερόμενος, όπως είπε η κυρία Ικονή ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Αλλά θα ήθελα να σας πω κυρίες και κύριοι ότι χρειάζεται και ρύθμιση, χρειάζεται και εποπτεία. Πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από την κρίση, να εξηγιάνουμε τα δημόσια οικονομικά διότι τα σημερινά χρέη θα είναι η φορολογία για τις επόμενες γενιές. Πρέπει να εξασφαλίσουμε καλή διακυβέρνηση και όλα αυτά δεν αρκούν. Χρειάζεται επίσης να υποστηρίξουμε ένα οικονομικό ε, πρόγραμμα όπως το είπα όπως το είπε χθες, το είπα και εγώ και το είπε χθες ο πρόεδρος Μπαρόζο και αυτό, αυτό το σκοπό θα έχουν οι προτάσεις μας του ε, φθινοπόρου για την ε, πράξη που θα αφορά την ενιαία αγορά διότι αν λειτουργεί αυτή η νέα αγορά καλύτερα θα είναι προς όφελος όλων μας και θα κλείσω με κάτι στο οποίο αναφερθήκατε πολλοί από εσά, ο συνάδελφος Ολυρέν και ο πρόεδρος Μπαρόσο ε, θα υποβάλουν σημαντικές προτάσεις για το θέμα της διακυβέρνησης στο τέλος του μήνα γιατί ο ευρωπαϊκό εξάμεινο στο οποίο αναφέρθηκαν πάρα πολλοί ομιλητές οπωσδήποτε πρέπει να δώσετε πολιτική όθηση σε αυτό το νέο σύστημα συντονισμού, ε, φωτογράφησης, προσδιορισμού ε, απέναντι στις κυβερνήσεις ενώ βεβαίως θα γίνονται σεβαστές οι αρμοδιότητες και οι προνομίες των εθνικών κοινοβουλίων εγώ όταν θα ψήφιζα το προπολογισμό της χώρας μου θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχής να γνώριζα να είχα μια εικόνα του τι γίνεται στις άλλες χώρες διότι μπορεί πολλές φορές με διαφορετικό τρόπο να καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα εάν εφαρμόζουμε μια πειθαρχία η οποία θα έχει συμφωνηθεί από κοινού. Ε, ε, σας διαβεβαιώ λοιπόν για τη βούληση και για την πρόθεση της Επιτροπής να προχωρήσει και να καταλήξει σε ουσιαστικά αποτελέσματα. Θα δώσω τώρα το λόγο στο Συμβούλιο, στον κύριο Ρέντε, μετά από τόσα συγχαρητήρια. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που χαιρετήσατε τη συμφωνία για την ε, χρηματοπιστωτική εποπτεία. Πολλοί θύμισαν ότι ήταν κοινή μα προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εισηγητών του, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Συμβουλίου. Πρέπει να σα πω ότι βρισκόμαστε στην αρχή μόνο τη διαδικασία. για να αποδείξουμε ότι η εποπτεία είναι ευρωπαϊκή υπεραξία και ίσω το πρώτο δίδαγμα που εξήχθη από τη χρηματοοικονομική κρίση θα πρέπει να επιλέξουμε ε, τα πρόσωπα με τον πιο αντικειμενικό τρόπο οι διαδικασίε βαίνουν προς την κατεύθυνση αυτή και επίση να αποδείξουμε και την αποτελεσματικότητα της εποπτείας στου διάφορους κλάδους. Αν θέλουμε όπω ζητήσατε πολύ, να προχωρήσουμε προς μία όλο και περισσότερο ευρωπαϊκή εποπτεία. Αποδεικνύοντας ε, ότι η συγκεκριμένη ε, συνδυασμένη και ολοκληρωμένη εποπτεία έχει νόημα ε, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Είναι όμως το πρώτο δίδαγμα και το πιο σημαντικό επαναλαμβάνω της κρίσης. Ε, θέσουμε τώρα τα θεμέλια για ένα νέο οικοδόμημα και σιγά σιγά θα ενισχύουμε τον πραγματικά ευρωπαϊκό χαρακτήρα της νέας αυτής μορφής εποπτείας. Επόμενο σχόλιο. Ο κύριος Γκοζές αναφέρθηκε σε αυτό προηγουμένως. Το απόγευμα θα εργαστούμε και πάλι στα πλαίσια ενός τριμερούς διαλόγου. Θα μιλήσουμε για τα επενδυτικά ταμεία θα πρέπει όλοι να κινηθούν, θα πρέπει όλοι να δεχθούν την ίδια πορεία με την υποπτία που μας επέτρεψε να επιτύχουμε. Είναι γεγονός ότι υπάρχει ακόμα εμπλοκή στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Ακόμα το συζητάτε αυτό ως προσωρισμένα στοιχεία ε, των επενδυτικών ταμείων, αλλά πρέπει να επιτευχθεί πρόοδος και εδώ. Και πιστεύω ότι συμφωνούμε τον κύριο Μπαρνιέ και επιθυμούμε να έχουμε ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα για τη θέση σε ισχύ των νέων κειμένων για τα επενδυτικά ταμεία. Θα προσπαθήσουμε ήδη από σήμερα να προχωρήσουμε, αλλά πρέπει έτσι κάπως να επιταχύνουμε, να έχουμε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό που να προστατεύει πραγματικά τους πολίτες και τους καταναλωτές στα πλαίσια ε, κάποιων προϊόντων ή δραστηριοτήτων που διεξάγονται διακινούνται στην επικράτεια της Ένωσης. Για να σας αναφέρω πώς έχει κατάσταση των πραγμάτων και συζήτηση, ο Μισελ Μπαρνιέ δήλωσε ότι στο άτυπο συμβούλιο θα γίνει μία σύγκριση, τι γίνεται κατέρωθεν του Ατλαντικού και εγώ προτίθεμαι να προσκαλέσω την πρόεδρο της Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής σας στο ΕΚΟΦΗΝ αυτό για να συζητήσουμε, να δούμε την πρόοδο των εργασιών. Αυτό δεν αφορά μόνο το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και το Κοινοβούλιο. Τέλει λοιπόν το μηνό θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και με το Κοινοβούλιο από αυτού του θέματο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να διαπιστώνουμε τι εξελίξει ε, και στην Ευρώπη. Επόμενο στοιχείο επιβολή κάποιου τέλους στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Ε, δεν θα επανέλθω στο Ταμείο Εξηγές που ενέφερε ο Μισελ Μπαρνιέ, ε, γιατί θα επανέλθουμε σε αυτό μέσα σε λίγες εβδομάδες. Δέκα χρόνια περίπου συζητούμε αυτό το θέμα. Στην προηγούμενη Βελγική Προεδρία του Συμβουλίου είχα προσπαθήσει να θέσω αυτό το θέμα στην μερίσια διάταξη προς αλλά δεν το καταφέραμε. Ήμασταν περίπου ομόφωνοι στο Βέλγιο και ήταν το μόνο θέμα στο οποίο ήμασταν ομόφωνοι τότε. Ε, τώρα, και δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό στο Βέλγιο, ναι. Τώρα η συζήτηση έχει ξεκινήσει, πραγματικά. Ακούω διάφορα αιτήματα έντονα για συγκεκριμένες προτάσεις για τους συντελεστές, τη φορολογική βάση και το πού θα πάνε τα έσοδα. Όλα αυτά καλά. Αλλά θα πρέπει να καταλαβούμε ότι σε κάποια ευρωπαϊκά κράτη αλλάζουν οι ιδέες και πρέπει να αλλάξουν για να ανοίξει πραγματικά η συζήτηση για τα πρακτικά δεδομένα για τους τρόπους. Για το G20, δεν παραπέμπουμε στο G20 το θέμα, αλλά προετοιμάζουμε το έδαφος για να δούμε με ποιους ε, εταίρους μας μπορούμε να πάμε στην ίδια κατεύθυνση. Θέλω να επιμείνω ότι θα συνεχιστεί με τρόπο ενεργό αυτή η συζήτηση. Έγινε ήδη στο ΕΚΟΦΗΝ χτες και τέλη ε, του μηνός το άτυπο ΕΚΟΦΗΝ θα συζητηθεί και είμαι προθυμός και θέλω πραγματικά να προχωρήσει η συζήτηση, ακόμα και για τη χρήση των πόρων. Βέβαια, ας μην γελιόμαστε, δεν μπορούμε να λύσουμε κρίσεις ή την κρίση μέσω αυτού. Μπορούμε να καταπολεμήσουμε την κερδοσκοπία και να βρούμε κάποιους πόρους που έχουμε ανάγκη και ε, ήδη τρεις με τέσσερις φορές θα μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Ε, κλιματική αλλαγή, αναπτυξιακή βοήθεια, να κλείσουμε τα ελλείμματα του προπολογισμού. καθένα βρίσκει και μία χρήση. Δεν θα είναι εύκολη λοιπόν η συζήτηση εκεί. Και Κύριε Πρόεδρε, τέλος θα ήθελα να μιλήσω και για την εξυγίαση των προϋπολογισμών, των ισοσκελισμών. Ας μην γελιόμαστε, το ευρωπαϊκό εξάμεινο είναι μία και μόνη φάση. Θα υπάρξουν και επόμενες, θα συζητήσουμε και για τις κυρώσεις. Τώρα οι προσανατολισμοί είναι να συζητήσουν πρώτα χώρε τη Ευρωζώνης μεταξύ του, και μετά θα δούμε πώ αυτό θα διευρυνθεί ε, και στα άλλα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δούμε τι λένε και που δεν είναι μέλη τη Ευρωζώνη. Η ιδέα είναι βεβαίως να έχουμε και μια μακροοικονομική σύγκληση με εξυγίαση των προϋπολογισμών μας, αλλά πρέπει να θυμίσω ότι το σύμφωνο που μας ενώνει είναι σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Ας μην ξεχνάμε το σκέλος της ανάπτυξης και τη συζήτηση για τις κοινωνικές πολιτικές, για την απασχόληση, για τις ε, περιβαλλοντικές πολιτικές. Δεν είναι το θέμα που μας απασχολεί αποκλειστικά να ισοσκελίσουμε τους προϋπολογισμούς μας. Όχι. Είναι και αυτό, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα προχωρήσουμε προς τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την κοινωνική πολιτική και την ενεργό συμμετοχή. Ενεργό, και το τονίζω, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Όλα αυτά, λοιπόν, είμαστε ε, σε μια φάση συζήτησης και η Βελγική Προεδρία ήδη από ε, σήμερα το απόγευμα θα το πράξει αυτό για τα επενδυτικά ταμεία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Προεδρεύον, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση αυτή και προχωρούμε στο επόμενο θέμα. Σύμφωνα με την ημέρα διάταξη, ακολουθεί η σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση. Έκθεση της κυρίας Γέγκλε, προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονική